Η δεύτερη ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλίας ε, κοινοποίησαν την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ζακ Κολομιέ από τις 2 Φεβρουαρίου 2018 η αντικατάσταση του κυρίου Εντουάρ Φέραν. ορίζω τον νέο συνάδελφο και υπενθυμίζω ότι καταλαμβάνει την θέση του και έχει όλα τα προνόμια και ασυλίες που ορίζει ο κανονισμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Έχετε κάτι επί της διαδικασίας? Ναι, γνωρίζω ότι συζητάμε, βλέπω εδώ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά δεν έχουμε συζητήσει το γεγονός ότι οι Βρετανοί συνεισφέρουν δισεκατομμύρια και θέλουμε τις συνεισφορές μας. Οπότε όλα αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ πέρα είναι